Καλησπέρα σας ε, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε λοιπόν. Εντάξει, δεν ξεκινάμε ακριβώς στις 7, διότι μερικοί συνάδελφοι είναι καθοδόν, ε, έρχονται, δεν ξέρω, με το λεωφορείο, με το τρένο, ε, με το αεροπλάνο, με τα πόδια. Λοιπόν, ε, ίσως να έχουμε αργήσει, καθυστερήσει λίγο, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε. Που σημαίνει ότι αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, η μερίσια διάταξη αυτής της έκτακτη συνεδρίαση μπορεί να εγκριθεί χωρίς καμία αλλαγή. Όσον αφορά στις ανακοινώσει μου, επειδή δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω, ε, θέλω δύο πράγματα να σας πω. Οι δύο βασικές επιτροπές, η Επιτροπή Προπολογισμών και η Επιτροπή ΕΚΟΝ, αποφάσισαν να ε, μεταφέρουν την ψηφοφορία για το FC2 στις 24 Απριλίου λόγω της πολιτικής σημασίας που έχει αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν για μας, για την Επιτροπή Ήτρε, ήταν απαραίτητο να προσαρμόσουμε και εμείς το πρόγραμμά μας, ε, να προσαρμόσουμε τη γνωμοδότησή μας και αναγκαστήκαμε να οργανώσουμε αυτή την έκτακτη ε, συνεδρίαση στο Στρασβούργο για να ψηφίσουμε για το FC2. Έχουμε δύο εκθέσεις. Η μία είναι νομοθετική και η άλλη είναι έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας και οι δύο είναι πολύ σημαντικές και θα θέλαμε να μεταφέρουμε την γνωμοδότησή μας και στις δύο επιτροπές, την Budget και την Econ, ε, γιατί έχουμε κοινή ευθύνη με βάση το, ε, τον κανόνα 65. Βασικά ενωνόμαστε με τις δύο αυτές επιτροπές με βάση το κανόνα 54, άρα δηλαδή για κάποια θέματα φέρουμε μεγάλη ευθύνη. Πάμε τώρα στο σημείο υπερθμών 3 της σημερινής διάταξης, έγκριση πρακτικών. Έχουμε τα πρακτικά της 28-29 Νοεμβρίου του 2016, της 12 Ιανουαρίου του 2017 και αν δεν έχετε κάποιο σχόλιο, θεωρώ ότι τα πρακτικά εγκρίνονται. Δεν υπάρχουν σχόλια. Περνάμε λοιπόν τώρα στην ε, ψηφοφορία. Έχουμε δύο προτάσεις ε, και πρώτα απ' όλα ε, να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσει η δοκιμαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Η ερώτηση ήταν αν σας αρέσουν οι ψηφοφορίες του Ρασφούγου. Έκλεισε η ψηφοφορία. Το κατάλαβα το μήνυμα, το πιασα. Πολύ σημαντικό μήνυμα. Ε, είχαμε και μία αποχή. Λοιπόν, ψηφίζουμε πρώτα για το σχέδιο γνωμοδότησης ε, σχετικά με τη νομοθετική πρόταση νέος κανονισμός ε, για ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως επίσης ε, και την εισαγωγή τεχνικών βελτιώσεων για το Investment Advisory Hub. Η συγγήτρια είναι η κυρία Καϊλή. Κύριε Πρόεδρε, μήπως μπορείτε να δείτε πώς είναι από το Αλκέτη, δεν έχω μαζί μου την κάρτα μου και θέλω να ξέρω αν μπορώ να ψηφίσω ή όχι. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Τροπολογία 114. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 115 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, αποδεκτή. Η 131 υπέρ, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Εσείς ψηφίσατε υπέρ, η κυρία Κουντίτσκα κατά. Δυστυχώς απορρίφθηκε όμως η τροπολογία. Ίσως να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα Άρα δηλαδή εγκρίνεται, εγκρίνεται η τροπολογία. Εντάξει. Εφόσον και εσείς είστε υπέρ, έχουμε δύο επιπρόσθετους υπέρ και έναν κατά. Ε, πρέπει να είστε πολύ υπομονητικοί. Εγώ ειλικρινά σας λέω, έχω μεγάλη υπομονή. Ένα, τρία, δύο υπέρ, κατά, αποχές, κατά. Ξανά. Ηλεκτρονική επανήλυση. Μάλλον θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε για την 132. Έκλεισε ψηφοφορία. Αποδεκτή. Η 17 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή. Η 18 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή. Η 134 μαζί με την 141 ή 134, κινούμε την 141 παρακαλώ. Ε, ψηφίζουμε και για τις δύο, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 19 υπέρ, κατά, αποχές, αποδεκτή. Η 135 υπέρ, κατά, αποχές, αποδεκτή. Η 144 υπέρ κατά αποχές. Αποδεκτή συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή. 138 υπέρ συμβαστική 2 Ελέγχουμε την ε, συμβαστική 2, κλείνει η ψηφοφορία, θα δούμε το αποτέλεσμα. Αποδεκτή. 138 υπέρ, κατά, αποχές, Κατανοώ ότι είστε κουρασμένοι, αλλά να σηκώνετε παρακαλώ το χέρι. 138 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 140 υπέρ κατά αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. 140 έκλειση ψηφοφορία. Άρα δηλαδή 28 προς 28 είναι το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. 1-4-2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Η 153, 153, δεύτερο τμήμα, η 153, δεύτερο τμήμα, υπέρ παρακαλώ, κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Ελέγχουμε την 153, το δεύτερο τμήμα της 153, κλείνει η ε, ψηφοφορία, απορρίπτεται. Η 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ κατά αποχές. Πάμε στη συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Συμβαστική 4. Ε, κλείνει η ψηφοφορία. Αποδεκτή. Η 100, μισό λεπτό, η 159, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 160, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 161, υπέρ, κατά, αποχές. 161, υπέρ παρακαλώ. Όχι, ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεν έπρεπε να πω υπέρ, έπρεπε να πω ηλεκτρονική επαλήθευση. Ζητώ συγγνώμη για την 161. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεν έχουμε πλειοψηφία. Άρα απορρίπτεται. 162. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 163. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή η συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή 181 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Θα πάρω. Θα κάνω δύο Αποδεκτή. Η 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 185 υπέρ τα αποχές απορρίπτεται, η 180 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 189 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση, ε, έκλειση ψηφοφορία, απορρίπτεται. Η 32 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβαστική 10. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική 11. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 193 υπέρ κατά αποχές, καλύτερα ηλεκτρονική επαλήθευση για την 193. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. γιατί είχαμε άλλη μία, μία επιπρόσθετη αρνητική ψήφο. 194 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ή 195 υπέρ, Η 196. Μισό λεπτό. Λοιπόν, 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται.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 καλύτερα να το ε, ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 204, τροπολογία 204, πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη, τροπολογία 205, υπέρ, κατά. Ίδια πλειοψηφία, επομένως απερίφθηκε η 205. 205. Ε, πέρας της Ναι, απερίφθη, απερίφθη. Τροπολογία 37. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 40. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβασμός 12. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 τμήμα 2 υπέρ κατά ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 46 τμήμα 2. 46 δεύτερο τμήμα λοιπόν, πέρας της ψηφοφορίας, απερίφθη. Συμβιβασμός 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 56, δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 56, δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 56, δεύτερο τμήμα. Πέρας της πληροφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 56, τμήμα 4. Τμήμα 4 λοιπόν της ίδιας τροπολογίας υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Αλλά καλύτερα να κάνουμε και μια επαλήθευση για την τροπολογία 56, τέταρτο το τμήμα, πέρας της ψηφοφορίας, γίνεται δεκτή. Τροπολογία 4, δεύτερο τμήμα. 4, δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά. Αποχές. Νομίζω πως γίνεται δεκτή, αλλά καλύτερα να κάνουμε μια επαλήθευση. Τροπολογία 4, τμήμα δεύτερο. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 63, δεύτερο τμήμα. Υπέρ Κατά. Ζητώ συγγνώμη που σας το λέω, αλλά έχετε το χέρι σας συνέχεια σηκωμένο και δεν καταλαβαίνω. Τροπολογία 63 δεύτερο τμήμα. 63 τμήμα δεύτερο. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 63, τρίτο τμήμα. 63, τμήμα τρίτο λοιπόν, υπέρ, κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Τρίτο τμήμα της τροπολογίας 63, πέρας της ψηφοφορίας και γίνεται δεκτό. Τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ, υπέρ 76. Να ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν επί της 76. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 88 υπέρ κατά αποχές απεριφθεί 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνθη 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 18 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση επί της συμβιβαστικής 18 άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας και εγκρίνεται τροπολογία 91 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 91. Πέρας. Δεκτή. 90 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 7 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 97. Πέρας της ψηφοφορίας, απερίφθη. Τροπολογία 99, υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 98, υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Συμβιβαστική 19, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 108 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απερίφθη ε, τελική ψηφοφορία διονομαστικής κλίσεως επί του συνόλου του ε, νομοθετικού ψηφίσματος και πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτό. Συγχαρητήρια κυρία Εύα Καϊλή. Προχωράμε λοιπόν στο επόμενο θέμα ε, που αφορά πάντα ε, την υλοποίηση της, ε, του ΕΦΣΥ. Είναι η εισηγητής ο Μαριάν Ζαν Μαρινέσκου πρώτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 35. Ελέγχουμε λοιπόν την τροπολογία 35 πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 τμήμα 2 22 τμήμα 2 υπέρ κατά αποχέσε ηλεκτρονική επαλήθευση. I close the vote. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές 54 υπέρ, κατά, δεκτό, 64 εγκρίνεται, 63 απορρίφτεται, 64 υπέρ, κατά, ας ελέγξουμε. 64, τροπολογία 64. Τέλος της ψηφοφορίας, απορρίπτεται, 65 υπέρ, κατά, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Υπάρχουν μικρές διαφορές, 65 Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε την 68 ε, πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε την 94 τροπολογία. Και πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά ας ελέγξουμε για την τροπολογία 113. 113. Πέρα της ψηφοφορίας 113 πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 114 υπέρ, κατά, αποχέσα, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τελική ψηφοφορία, ονομαστική, άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα πέρα της ψηφοφορίας Έχουμε πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον ε, εισηγητή. Τέλος ε, με το ε, θέμα 4. Έχετε στα διάφορα κανένα θέμα πέρα της ψηφοφορίας.